Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Benvenuti a tutti. Καλώς ορίσατε. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη καταρχάς και να ζητήσω συγγνώμη για αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Ευθύνη των συντονιστών. Εγκρίνουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Είχαμε προβλέψει να είναι εδώ ο Υπουργό Σάιμον Κόβενι, πρώην ε, ε, Προεδρεύων του Συμβουλίου, για να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της Ιρλανδικής Προεδρίας, αλλά μας ενημέρωσαν ότι σήμερα και αύριο ο Υπουργό πρέπει να βρίσκεται στην Ιρλανδία για επίγοντα ζητήματα. Επομένως, ο Υπουργός ε, μου ζήτησε να σας διαβιβάσω την λύπη του, διότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στην συνεδρίασή μας, αλλά είναι διατεθειμένος ε, για να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων το Σεπτέμβριο. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν κάποιες άλλες προσθήκες, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με αυτή την αλλαγή. Να σας πω επίσης ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου και υπάρχει δυνατότητα διερμηνίας σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Σημείο υπαριθμών 4. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 29ης και 30ης Μαΐου. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά. Και να περάσουμε τώρα στο σημείο 5. Δημιουργία δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης όσον αφορά τα εισοδήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο εισηγητής είναι ο Τζανκάρλος Κοτά και θα ψηφίσουμε το ενοποιημένο κείμενο του κανονισμού για την οικονομία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας υπενθυμίσω ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα ευθυγράμμισης και ο κύριος Σκοτά στη συνεδρίαση της 31ης Μαΐου μας εξέθεσε τις απόψεις του και έχουμε ψηφίσει. Εγκρίθηκαν 31 τροπολογίες, καθώς επίσης και αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Να σας υπενθυμίσω ότι έγινε και ένας πρώτος τριμερής διάλογος, επομένως υπήρξαν και αρκετέ τεχνικές συνεδριάσεις και οι ημερομηνίε ήταν 24 Ιανουαρίου, 9 Απριλίου και ούτω καθεξής. Στο κείμενο λοιπόν που έχουμε ενώπιόν μας έχουμε τις αλλαγές οι οποίες προέκυψαν από αυτές τις τεχνικές συνεδριάσεις και είναι το κείμενο το οποίο ενέκρινε ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές μετά από τις διαπραγματεύσεις. Εάν θέλει το λόγο ο εισηγητής να τον δώσω, αλλιώς θα περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Θέλετε το λόγο? Όχι. Ο κύριος Άγνιου θέλει κάτι διαδικαστικό. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα δίλημα. Έχω αφήσει την κάρτα ψηφοφορία μου στο μηχάνημα στο Στρασβούργο. Ή θα ψηφίσουμε χωρί ηλεκτρονικέ κάρτε, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα, ή θα επιμείνετε, επομένω θα πρέπει να πάω να τη φέρω. Αλλά μέχρι να επιστρέψω μπορεί να έχει τελειώσει και ψηφοφορία. Τι να κάνω. Μην ανησυχείτε, θα το ρυθμίσω εγώ. Η Ράτσα θέλει το λόγιο. Κύριε Γκαρθία Πέρες. Το ίδιο κι εγώ. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορείτε να με καταμετρήσετε και εμένα. Ωραία. Bene, allora voto aperto. Si va... Άρχεται η ψηφοφορία, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Άγνιου και η κυρία Γκαρθία Πέρες δεν έχουν ε, κάρτες, επομένως σας παρακαλώ διανατάσσεως χειρός να εκφράσετε την άποψή σας, μόνο για σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπέρ, κατά κύριε Άγνιου. Απέχει ο κύριος Άγνιου και κατά η Ράτσα. Πέρασε της ψηφοφορίας. Μισό λεπτό. Ο Μάρκ υπερψηφίζει ή ψηφίζει κατά. Ωραία. Ωραία. Εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ, 8 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Σκοτά. Ο κύριος Ταραμπέλα. Για ενημέρωση και μόνο κύριε Πρόεδρε, για να μην δοθεί εντύπωση ότι όπως θέλει ο κύριος Άκνιου ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός δεν λειτουργεί και υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελών υπάρχει μια δεύτερη κάρτα. Εάν ξεχάσετε λοιπόν την κάρτα της υπάρχει γραφείο δίπλα στον Ολομέλεια, υπάρχει και μια κυρία υπεύθυνη, κυρία Πορτέλα αν δεν κάνω λάθο, μπορείτε κάλλιστα να πάτε να τη βρείτε, έχει κάρτα και θα σας περιμένει να σας τη δώσει. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση Μάρκ. Ωραία. Να περάσουμε στο σημείο 6. Σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Καθεστώς συναλλαγών που εφαρμόζονται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταπίεση γεωργικών προϊόντων. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, ο υποφαινόμενος είναι ο εισογητής για την έκθεση αυτή. Και πέραν των εννέων τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης, λίγο ησυχία παρακαλώ, προσοχή. Έλεγα λοιπόν, όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι συγγετής για την έκθεση αυτή. Πέραν των εννέα τροπολογιών στο σχέδιο έκθεσης, τα μέλη της Επιτροπής μας υπέβαλαν επιπλέον έξι τροπολογίες. Και υπάρχει και μία γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, της οποίας συντάκτης ήταν ο συνάδελφος ε, Άλβερ Ντένς. Ε, στην γνωμοδότηση αυτή είχαμε ακόμα 12 τροπολογίες. Βάσει της πολιτικής συμφωνίας ε, στην οποία καταλήξαμε για την ενιαία ΚΟΑ, θα ήθελα να ζητήσω να αποσυρθούν οι τροπολογίες 1 και 7 του εισηγητή. Πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες ε, αφορούν το άρθρο 43 σημείο 3, στο οποίο σε επίπεδο ΚΟΑ με την ε, έκθεση Αρτέν εγκρίναμε ήδη μια συγκεκριμένη συμφωνία. Έχουμε καταλήξει σε τελείως διαφορετική συμφωνία και για λόγους συνοχής λοιπόν με αυτή τη συμφωνία θα ήθελα να ζητήσω να αποσυρθούν οι τροπολογίες 1 και 7. Θα ήθελα να σας επισημάνω επίσης ε, και ένα αίτημα για κατατμήματα ψηφοφορία το οποίο έκανε η κυρία Αγιούζο για την τροπολογία 8 της Επιτροπής ΙΝΤΑ και ζητά λοιπόν να ε, ε, γίνει κατά τμήματα ψηφοφορία για τη φράση «ο ελ πούμπλικο». Κύριε Ντές, θέλετε να λάβετε το λόγο. Αν όχι, μπορούμε να ψηφίσουμε απευθεία. Ωραία, ψηφίσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση λαμβάνουμε υπόψη και την ψήφο του κυρίου Άγνιου. Να ξεκινήσουμε μόλον διανατάσσεως χειρός, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα για τις κάρτες. Υπέρ. Είναι τα τρία. Υπέρ. Κατά. Διανατάσσεως χειρός. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι τα 6 υπέρ, υπέρ της είναι τα 6 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε να κάνουμε επαλήθευση. Ωραία. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την ίντα 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, και ε, η Πέραση ψηφοφορία. What is it? Εγκρίνεται. Ήταν 15-15 με ε, την, ψήφο τη θετική του κ. Άκλου Εγκρίνεται η ΙΝΤΑ 6. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 3 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 Γιούζο υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Είναι τα 7 υπέρ. Επαλήθευση λοιπόν για την 14 γιουζο. Άρχεται η ψηφοφορία. Σημειώστε επίσης ότι ο κύριος Άγνιου είναι υπέρ. και η Ράτσε κατά. Παρακαλώ. Με χτύπησε ο ήλιος και ψήφισα λάθος. Θέλω να αλλάξω την ψήφο μου σε θετική για να συνάδει και με την άποψη της ομάδας. Τι να κάνω, το παραδέχομαι. Δεν είναι αργά, προλαβαίνω. Συνάδελφοι, να ψηφίσουμε και πάλι σας παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία για την ε, τροπολογία 14 Αγιούζο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο μόνο ψήφους, μία υπέρ και μία κατά. 15-15 απορρίπτεται λοιπόν. Είναι τα 7 ο χειρό, Υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Στην ίντα 8 πρέπει να ψηφίσουμε κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 9. Υπάρχει και μια προφορική τροπολογία για αλλαγή από 5 σε 7 χρόνια. Προσοχή λίγο λοιπόν. Στην τροπολογία 9 υπάρχει και μια προφορική τροπολογία και εδώ και πάλι για να συμμορφωθούμε στη συμφωνία που επιτύχαμε για την ΚΟΑ, σας το λέω στα αγγλικά, shall be confirmed the Commission for a period of 7 years from και όχι 5 years που είχαμε πριν. Συμφωνείτε, τη δέχεστε, ευχαριστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Ίντα 10 υπέρ. Για την Ίντα 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ίντα 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Και τέλος είναι τα 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, Ίντα 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα δύο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της νομοθετικής πρότασης ως τροποποιήθηκε υπέρ, α, συγγνώμη, ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζουμε πάντα ότι έχουμε και τις ψήφους του κυρίων Άκνιου και της κυρίας Γκαρθία Πέρες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Απέχει ο κύριος Άγνιου. Εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ. Και τώρα ψηφίζουμε και πάλι ηλεκτρονικά για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. Ευχαριστώ. Και τέλος, μια τελευταία ψηφοφορία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο με στόχο συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και μια αποχή. Ωραία. Πολύ μεγάλη πλειοψηφία. 30 ψήφοι υπέρ. Σας ευχαριστώ όλους. Ολοκληρώθηκε και το σημείο αυτό. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι ψηφοφορίες. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Προσέξτε τώρα, στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης δεν θα πρέπει να σας ε, τυχαίει ο τίτλος που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, διότι το θέμα που συζητάμε τώρα αφορά τους μεταβατικούς κανόνες για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής εν γέννη. Και έχουμε το κείμενο για τους μεταβατικούς κανόνες. Η πρώτη συζήτηση που γίνεται στην ε, ε, Επιτροπή μα για του μεταβατικού αυτού κανόνε, Εισηγητής είναι ο κύριο Ντε. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι περιλαμβάνονται στοιχεία για τι Νομοθετικέ διαδικασίε για την κοινή γεωργική πολιτική, τα οποία βρίσκονται ακόμα εντό παρενθέσεων στο κείμενο το οποίο έχουμε συζητήσει με την Ιρλανδική Προεδρία. Πρόκειται λοιπόν για τα σημεία τα οποία συζητήσαμε προηγουμένω στη συνεδρίαση των συντονιστών και ακόμα είμαστε στη διαδικασία τη διαπραγμάτευση για τα σημεία αυτά. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον Άλμπερτ και να του δώσουμε τη δυνατότητα να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Έχεις το λόγο, Άλπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως μόλις είπε ο Πρόεδρος, στην συνάντηση των συντονιστών ήδη παρουσίασα Κάποια από αυτά που συζητούμε εδώ πρόκειται για την πρόταση της Επιτροπής. Έχουμε και τις ε, ιδέες ε, του Συμβουλίου και δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε. Πρόκειται για μια πολύ τεχνική έκθεση, μια δύσκολη επί της έκθεση, γιατί βασίζεται σε πολλές άλλες οδηγίες και πολλούς άλλους κανονισμούς. Και εδώ καλούμε, καλό εμείς να συγκεντρώσουμε όλες ε, τις ιδέες αυτών των οδηγιών και κανονισμών. Θα ήθελα να σας πω το συντομότερο δυνατό να μου υποβάλλετε τροπολογίες. Ζητώ από όλους τους συναδέλφους να έρθουν σε επαφή με τις κυβερνήσεις τους έτσι ώστε οι επιθυμίες και οι προτάσεις να μπορέσουν να ενσωματωθούν ομαλά στο κείμενο της έκθεσης. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε έτσι ώστε να γίνει με ομαλό τρόπο η μετάβαση στα νέα προγράμματα, γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση. Είτε θα πρέπει λοιπόν να επιμικίνουμε την ισχύ των παλιών κανόνων έτσι ώστε να περάσουμε ομαλά προς τους νέους κανόνες και τη νέα χρηματοδότηση γιατί αν δεν εγκριθεί η μεταβατική αυτή περίοδο με ομαλό τρόπο κινδυνεύουμε να έχουμε διακοπές και ε, διαταραχές. Θα είναι προβληματική η συνέχεια αν δεν αποφασίσουμε εκ των προτέρων πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση από τους παλιούς τους καινούριους κανόνες. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν να με ενημερώσετε πώς βλέπετε και πώς βλέπουν οι κυβερνήσεις σας ε, την συνέχεια Επίσης, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε τι θα γίνει σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 14 κράτη η κατάσταση προϋποθέτει νέες επενδύσεις αν θέλουμε να συνεχιστούν τα προγράμματα. Θα ήταν λογικό λοιπόν για το 2014 να προβλέψουμε τι θα γίνει όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις. Επίσης Επιτροπή προτείνει να αλλάξουν κάποιοι κανόνες όσον αφορά το χρόνο που διαθέτουν τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή σήμερα προτείνει 7 ημέρες. Ε, αυτό δεν είναι αρκετό. Εγώ προτείνω τουλάχιστον 3 μήνες, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και έτσι ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να πάρουν αποφάσεις. Δεν μπορεί ένα κρατός να αποφασίσει μέσα σε μία εβδομάδα ιδιαίτερα όταν ε, υπάρχει Συμβούλιο Υπουργών, παραδείγματος χάρη. Εγώ προτείνω λοιπόν οι 7 ημέρες να ε, μετατραπούν σε 3 μήνες. Έχουμε συζητήσει επίσης και το ξανασυζητήσαμε εδώ στους συντονιστές το θέμα των μεταφορών των ε, ποσών. Όπως προτείνει η Επιτροπή και το θέμα αυτό συζητείται εδώ και αρκετό καιρό, οι μεταφορές από την πρώτο πυλώνα στο δεύτερο πυλώνα ή από το δεύτερο στον πρώτο. Η Επιτροπή, επαναλαμβάνω εδώ, έχει δώσει τη δυνατότητα σε κάποια κράτη-μέλη να μεταφέρουν από, τη δεύτερη, από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Υπάρχουν, αν θέλετε, κράτη-μέλη που έχουν ε, πολύ ψηλά ποσοστά κονδυλίων στο δεύτερο πυλώνα και λογικά θα πρέπει η μεταφορά ποσών από το δεύτερο στον πρώτο να μπορεί να γίνουν. Μέχρι τώρα βεβαίως προβλέπεται μόνο το 7% των κονδυλίων να μπορεί να μεταφερθεί, αλλά μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Η Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη, η οποία έχει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό στο δεύτερο και πολύ χαμηλό στον πρώτο πυλώνα, σε αυτή την περίπτωση για το 2014 θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα σε αυτό το κράτος και σε άλλοι να μεταφέρουν τα ποσά από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Ελπίζω αυτές οι προτάσεις και άλλες να υποστηριχθούν έτσι ώστε να γίνουν κάποιες, ε, να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε κάποια ποσά και να τα χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο. Τώρα, από το 2014 και πέρα, δίνονται δυνατότητες, οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να προαποφασιστούν ποια είναι τα ποσά που μπορούν και πρέπει να μεταφερθούν. Από το 2013 στο το 2017 θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες για διορθώσεις υπάρχουν. Αυτό μου φαίνεται λογικό από τη στιγμή βεβαίως που θα γίνει μια γενικότερη αξιολόγηση των αναγκών χρηματοδότησης. Μέχρι το 2017 λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μία παράταση σε κάποια κράτη-μέλη και την ίδια ώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε κανόνες ε, από σήμερα μέχρι το 2017. Δεν είμαι τελείως σίγουρος αν αυτό θα αποφασιστεί, αλλά εγώ τουλάχιστον το θεωρώ σαν απαραίτητο, σαν αναγκαίο. Πιστεύω επίσης ότι όλοι συμφωνείτε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να γίνει σταδιακά. Δηλαδή μια πρώτη φάση της αγροτικής μεταρρύθμισης το 2015 όσον αφορά την λεγόμενη εξωτερική σύγκληση. Αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από το 2014 και η εξωτερική σύγκληση για τα κράτη που εμπλέκονται είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκινήσει ήδη από το 2014 για να προετοιμαστεί το 2015. Εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Πριν ε, τις ε, καλοκαιρινές διακοπές, εγώ θα έχω έτοιμο το κείμενό μου. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο και θα το δώσω για μετάφραση. Και ελπίζω το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά για να είμαι πιο ρεαλιστή, θα σας έλεγα τέλος Σεπτεμβρίου θα είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Αυτά. Πολύ καλά, ευχαριστούμε Άλμπερτ. Ακούσαμε λοιπόν μια παρουσίαση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού θέματος για τους μεταβατικούς κανόνες. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν θα πρέπει να σας εγχαίει ο τίτλος στο σημείο της σημερινής διάταξης. Το θέμα αφορά τους μεταβατικούς κανόνες για όλο το θέμα της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε με τις παρεμβάσεις. Ο Ερικ Αντριέ, Κόστινζερ και η Λυπή. Ερικ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Άλμπερτ για την παρουσίαση της έκθεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και λεπτό θέμα γιατί φυσικά αφορά πάρα πολλά κράτη-μέλη που όπως είπες πολύ σωστά έχουν ε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να γίνει με ομαλό τρόπο αυτή η μετάβαση από τον παλιό στο νέο κανονισμό τα παλιά προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέα κονδύλια, με νέα χρηματοδότηση και από το 2015 και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσει η χρηματοδότηση και η προσαρμογή των προγραμμάτων. Τελικά όλοι θα πρέπει να έχουμε τον ίδιο στόχο, δηλαδή μια εγγύηση, μια σταθερότητα και νομική ασφάλεια γιατί δεν είναι δυνατόν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να συνεχίζουν αν δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι ακριβώς το πλαίσιο για το μέλλον. Η πρόταση λοιπόν της Επιτροπής φυσικά είναι ανεπαρκής. Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής πριν από 7 χρόνια είχε παρόμοια προβλήματα, βρέθηκε μία λύση, μία λύση προβληματική θα έλεγα για την ε, μεταβατική περίοδο και είδαμε ότι δεν αρκεί η πρόταση της Επιτροπής. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξανακάνουμε το ίδιο. Πάρα πολλοί ε, επικεφαλής ε, αγροτικών εκμεταλλεύσεων φοβούνται σήμερα ότι θα βρεθούν σε μια παρόμοια κατάσταση. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για αυτούς οι οποίοι είναι κτηνοτρόφοι και περιμένουν αυτές τις επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί πολύ συγκεκριμένη λύση για αυτή τη μεταβατική περίοδο. Το ίδιο θα έλεγα και για τις άμεσες πληρωμές. Πρέπει να βρούμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει και το οποίο θα ικανοποιεί τους ενδιαφερόμενους. Ίσως μια λύση θα ήταν τα κράτη-μέλη να αναλάβουν αν θέλετε αυτές τις ε, πληρωμές βάσει πολύ συγκεκριμένων κριτηρίων βεβαίως για αυτό το συγκεκριμένο έτος έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες να κινηθούν. Αυτό μπορεί να είναι μια λύση, μια δυνατότητα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Μακάρι τέλος Σεπτεμβρίου να είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε. Επαναλαμβάνω, το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσθέσουμε αβεβαιότητα και ασάφεια στον γεωργικό τομέα. Επαναλαμβάνω και εγώ αυτό που είπε Άλμπερτ, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε συγκεκριμένες ενδείξεις και να τις στηρίσουμε για αυτό το μεταβατικό έτος. Το συντομότερο δυνατόν λοιπόν θα πρέπει να ψηφίσουμε και να προτείνουμε μία ε, λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Έρικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή δεν είχαμε γραπτή ε, θέση, τοποθέτηση του Αλμπερντές ε, είναι ανάμεσα στην έκθεση 7 και στην 9 και νομίζω ότι όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με τον προϋπολογισμό επίσης. Συνεπώς εγώ έλαβα γνώση των προτάσεων της Επιτροπής και θα περιοριστώ στο να κάνω μια εκτίμηση ε, σχετικά με τις προτάσεις αυτές. Ε, σχετικά με την γενική ανάλυση, έχουμε ξεκινήσει από την μεταρρύθμιση που αναφέρεται στην αγροτική ανάπτυξη και οι οριζόντιοι κανόνες ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα εφαρμοστούν στο ακέραιο. Δεν ισχύει το ίδιο για τις άμεσες πληρωμές που είναι ό,τι βαθύτερο έχουμε για την μεταρρύθμιση. Η άμεση υποστήριξη θα γίνει με μια διαφορά χρονική για να προετοιμαστούν καλύτερα τα πνεύματα των αγροτών και η λειτουργία των δικήσεων για τις βασικότερες αλλαγές και αυτό είναι ακρογωνίας λήθος της μεταρρύθμισης. Στις διάφορες συναντήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους του επαγγέλματος στις χώρες μας, είδαμε ότι περιμένουν ε, με ανυπομονησία αυτή τη μεταρρύθμιση. Οι αγρότες θέλουν να βρουν προοπτικές και πολλοί πολίτες επίσης επιθυμούν η δημόσια αγροτική πολιτική να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες τους. Σήμερα βρέθηκε ένα συμβιβασμός και αν δεν είναι το ιδανικό το οποίο θα ήθελα, επιτρέπει να υπάρξουν, να υλοποιηθούν σημαντικές αλλαγές και ε, χαιρετίζω την ε, εικόνα που δόθηκε για να κλείσουν ε, οι τριμερείς διάλογοι της Ιρλανδικής Προεδρίας και θα πρέπει τώρα να συγκεκριμενοποιήσουμε τα πράγματα και με την αυξανόμενο ευροσκεπτικισμό θα πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρώπη δρά έχει πράξεις, δράσεις και από αυτό εξαρτάται η δημόσια αξιοπιστίες μας θα ήθελα διάφορα μέτρα να τα σε αυτό το στόχο. Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, θα πρέπει να μπορέσουμε να διευρύνουμε την ταχεία εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης σε ορισμένα στοιχεία της ρύθμισης, κυρίως σε αυτά που προϋπήρχαν στην σημερινή λειτουργία της κοινή αγροτικής πολιτικής και για τα οποία η υλοποίηση εφαρμογή είναι σχετικά απλή από διοικητικής απόψεως και αναφέρομαι κυρίως τους νέους κανόνες για την αποσύνδεση όπου μόνο ε, οι συντελεστές σύζευξης, σύνδεσης έχουν κάπως τροποποιηθεί. Επίσης σκέφτομαι την ανανέωση των εθνικών ενισχύσεων που επιτρέπονται σε ορισμένε χώρες συμπληρώνοντας τις κοινοτικέ άμεσες ενισχύσεις. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα πρέπει ε, ήδη από το 2014 να ισχύσουν. Όσον αφορά τον τομέα των άμεσων ενισχύσεων, τα μέτρα, τα μεταβατικά αναφέρονται στην προσαρμογή εφαρμογή των επιπέδων στήριξης και όλων των υποκειμένων ε, μηχανισμών ε, σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι ε, μειώσεις της Κομισιόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται γραμμικά σε όλες τις πληρωμές της κίνησης ΚΑΠ, ούτως ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμού για τα κράτη-μέλη, όπως αυτά που υποστηρίξαμε στην μεταρρύθμιση για την ανακατανομή ε, των ενισχύσεων. Τέλος, όσον αφορά την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο τη μεταβατική 2014, η Κομισιό προτείνει ανανέωση μόνο ενός μέρους των ενισχύσεων που σχετίζονται με την επιφάνεια ε, και ανάλογα με το εισόδημα, το ετήσιο των δικαιούχων ε, πληρωμές Natura 2000 και άλλες και στα πλαίσια της ε, οδηγίας πλαίσιο για το είδωρ. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για τα άλλα μέτρα. Τα κράτη-μέλη ε, μπορούν ε, να τα περιλάβουν στις δεσμεύσεις τους χωρίς να είναι βέβαιοι ότι θα εγκριθούν στον επόμενο προγραμματισμό τους και στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος να μην γίνουν επιστροφές για το μέρος της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης και θα ήθελα να προτείνω δύο προτάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Ή θα πρέπει να, να διευρύνουμε τον κατάλογο των μέτρων που θα περιληφθούν ε, στην ισχύουσα ρύθμιση και κυρίως ε, την στήριξη για την εγκατάσταση και για τις επενδύσεις ε, που τροποποιήθηκαν από τη μεταρρύθμιση ή απλώς θα πρέπει να παρατείνουμε για ένα έτος μέχρι τέλους 2014 τον συνεριμερινο προγραμματισμο προγραμματισμό 2017-2013, ούτως ώστε να εξαλειφθεί κάθε αβεβαιότητα νομική και οικονομική ως ε, προς ε, την ε, πληρωμή και να μην φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν αν δεν εφαρμόσουν τα μέτρα το 2014. Αυτή η αναχρονιστική κατάσταση θα ήταν πολύ επιζήμια ε, για τους υποψήφιους για εγκατάσταση και για αυτούς που θέλουν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Αυτό το κενό θα είναι επιζήμιο για την εικόνα της Ευρώπης. Ευχαριστώ, Ερίκ. Ο Τζόρτζ Λάιον και μετά ο Κάπουλα Σάντο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Άλμπερτ, για αυτήν την ενημέρωση και νομίζω ότι από την άποψη της νέας ΚΑΠ είναι χρήσιμο να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τα νέα προγράμματα στα να δώσουν την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν έναν προγραμματισμό που θα ισχύσει το ε, συντεμότερο δυνατόν. Ε, νομίζω ότι 2015 θα πρέπει να περιμένουμε και τις άμεσες ε, πληρωμές. Αν δούμε τον αριθμό των κατεξουσιοδότηση πράξεων, ίσως θα πρέπει να περιμένουμε τον Νοέμβριο για την εφαρμογή, την υλοποίηση των πληρωμών αυτών με λεπτομέρειες. Ένας τομέας που θα θέλετε να εξετάσετε είναι η ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Βεβαίως θα θέλαμε να αλλάξει και σχέση με τη νέα συμφωνία ε, το όριο αυτό, ποιος ε, τηρεί την πειθαρχία και ποιος δεν την τηρεί. Όσο προς τους πυλώνες, νομίζω ότι αναφέρατε την θέση ε, της, ε, του Κοινοβουλίου σχετικά με τις άμεσες ε, πληρωμές και το πακέτο. Δεν χρειάζεται να έχουμε δύο χωριστές αποφάσεις, μια που διαπραγματευόμαστε και την άλλη και το πακέτο που εσείς εκπονείτε. Θα πρέπει να έχουμε συνεκτικότητα στην όλη προσέγγιση για να επιτρέψουμε στις διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο Λουίς και μετά ο Φέιμο. Ε, ε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα επί τη ευκαιρία να πω στον Άλμπερτες ότι θα συνεργαστώ μαζί του προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εκκρεμούν ακόμα στη διαπραγμάτευση ε, μετά το τέλος της ελληνικής Προεδρίας και πάντα λέγαμε ότι πρέπει να διαπραγματεύσουμε όλα τα κεφάλαια της ε, ΚΑΠ, αλλά αυτή την ερμηνεία δεν την ασπάστηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τελικά πίστηκαν και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ε, σημεία τα οποία κρεμούν, τα οποία ε, αφορούν και το μεταβατικό κανονισμό. Ε, οι μεταφορές ε, που αναφέρθηκαν από τον Άλμπερντες. Ναι, σίγουρα πρέπει να κάνουμε κάτι, διότι ε, ερίζουν οι απόψεις μεταξύ ημών και του Συμβουλίου. Το 5% που πρέπει να περάσει από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα, ναι μεν θα μπορούσε να μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μεταφορά από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Και η θέση του Συμβουλίου είναι πολύ αυστηρή και το περιθώριο ευελιξία είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Θα πρέπει λοιπόν να διαπραγματευτούμε όλες αυτές τις ε, πτυχές, αλλά και με τρόπο ώστε να τιμούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να προσυπογράφουμε ό,τι αποφασίζει το Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι απαρνόμαστε την ε, συναπόφαση και απλώς ε, δεχόμαστε ό,τι μας λένε. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα διαπραγματευτούμε από το Σεπτέμβριο, όπως είπα και στους συντονιστές, ε, θα παρουσιάσω κάποιες συμβιβαστικές προτάσεις και θα δω με τους κοιόδους συζητητές πώς μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη συμφωνία εδώ, στο Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και αυτή τη συμπεφωνημένη θέση μας στο Συμβούλιο, για να διαπραγματευτούμε μια συνολική συμφωνία, για να την εγκρίνουμε στη συνέχεια και στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Είναι σαφές ότι πολλές από αυτές τις πτυχές της διαπραγμάτευσης έχουν σχέση και με την έκθεση του κυρίου Ντές, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συντονιστούμε για να ε, μπορέσουμε να έχουμε τα καλά αποτελέσματα που θέλουμε. Ο κύριος Φέιμον και μετά η Μπρίτε Ρέιμαρς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική νομοθεσία και βεβαίως ε, αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε εδώ είναι τι θα γίνει το 2014. Πρέπει να βρούμε μία λύση, ένα συμβιβασμό που να μας επιτρέπει να μην χαθεί το έτος 2014, να μην είναι έτος απώλειας για τους ε, αγρότες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναβάλουμε ή να καθυστερήσουμε γιατί αυτό θα έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες και απώλειες για τους ε, γεωργούς. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι στην έκθεση αυτή να δώσουμε περισσότερη ευελιξία στα κράτη-μέλη έτσι ώστε για το 2014 να μπορέσουν τα κράτη-μέλη μέσα κονδύλια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό να τα χρησιμοποιήσουν και να συνυπολογιστούν. Βεβαίως ε, και εμείς θα κάνουμε κάποιες προτάσεις που θα συζητηθούν πιστεύω στα πλαίσια των τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ Μπρίτα Ρέμερς. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Ναι, θα υποβάλουμε τροπολογίες. Ο Άλμπερτ μίλησε για προηγούμενες οδηγίες και κανονισμούς. Ήδη όμως έχουμε συμφωνήσει σε πολλά από αυτά με το Συμβούλιο στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που είχαμε. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Την τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι προτείνουμε για τα μεταβατικά μέτρα. Η τελική ψηφοφορία βεβαίως στοχεύει στην αγροτική μεταρρύθμιση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μεταβατικό ε, τμήμα των μέτρων και βάσει αυτού θα πρέπει να αποφασίσουμε. Χαίρομαι γιατί πιστεύω ότι θα ακολουθήσει μια πάρα πολύ ζωντανή συζήτηση. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι για να λάβουν το λόγο. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο και πάλι στον εισηγητή, στον Τέσ, να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη, εάν θέλει φυσικά. Είστε εδώ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ναι, ε, βεβαίως χρειάζεται αυτή η πρόταση, θα πρέπει από το τέλος του έτους να υιοθετηθεί για να έχουμε μια βεβαιότητα ε, σχετικά με το τι θα συμβεί για τις ενισχύσεις για τους αγρότες και να ξέρουμε επίσης τι θα συμβεί με την δίκηση στο 2014. Θα περιοριστώ σε τρία σημεία. Πρώτον, όσον αφορά τα διάφορα στοιχεία και την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων, της πληρωμές, το πολιετές πλαίσιο, ε, περαμένουμε ε, βεβαίως ε, δεν έχουμε ακόμα συμπεράσματα ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για το πολιετές πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβιολία ότι ε, τι θα, πώς θα είναι αυτά τα στοιχεία από την άποψη της μεταρρύθμισης και εδώ στην ρύθμιση την μεταβατική θα πρέπει να προσαρμοστούν καταλήλως ε, για να έχουμε την ίδια διατύπωση αλλά και τα δύο στοιχεία υπάρχουν στην πρότασή μας η εξωτερική σύγκληση και η ευελιξία ανάμεσα στους πυλώνες. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αγροτική ανάπτυξη. Το γεγονός ότι προτείναμε την δυνατότητα ε, να, να, έχουμε ε, στοιχεία ε, για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης με νέα κονδύλια. Τα μέτρα αυτά είναι συνδεδεμένα με την εφαρμογή των άμεσων πληρωμών από την δίκηση. Τα δύο πάνε μαζί, οι αγρότες κάνουν την αίτησή τους ταυτόχρονα και για τις άμεσες πληρωμές και για την αγροτική ανάπτυξη. Γι' αυτό έχουμε εδώ προβλέψει ειδικού κανόνες για όλα τα άλλα στοιχεία δεν βλέπουμε καμία ανάγκη να υπάρχει ε, ιδιαίτερη μεταβατική μεταχείριση σε αυτούς τους τομείς. Ο προγραμματισμός για τη νέα περίοδο θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης να υλοποιηθούν τα μέτρα το σύντομότερο δυνατόν. Αν συγκρίνω με τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία, εκεί δεν υπάρχουν ρυθμίσει μεταβατικές. Είναι φυσικό τα νέα κονδύλια να ξοδευθούν για τα νέα προγράμματα. Αυτά θα πρέπει να είναι οι κανόνε, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε την μεταρρύθμιση την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε ειδικά μέτρα να ακολουθήσουν την λογική των άμεσων πληρωμών και γι' αυτό θα πρέπει στο πλαίσιο αυτής της πρότασης να ληφθούν υπόψη ξεχωριστά. Για το θέμα του ίνου και της ζάχαρης δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη ειδική μεταχείρισης ή μεταβατικοί κανόνες σε αυτών των κανονισμών. Υπήρξε πολιτική συμφωνία στα πλαίσια της μεταρρύθμισης και αυτή η πολιτική ε, συμφωνία θα ενσωματωθεί στην ρύθμιση που συζητήσαμε τον Ιούνιο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται εδώ να προσθέσουμε κάτι για την μεταβατική περίοδο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ωραία. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Αλμπερντές, θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω τους φίλους από την αντιπροσωπεία της Ελίζαμπεθ Γέγκελ που είναι εδώ και παρακολουθούν ε, τη συνεδρίασή μας. Ε, είναι όλοι εκ Γερμανία. Τους καλωσορίζουμε και τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Να δώσω το λόγο στην Ελίζαμπετ για να τους καλωσορίσει και από εκεί και πέρα στον Άλμπερντ Ντέσ για να ολοκληρώσουμε. Ελίζαμπετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί τους χαιρέτησα, τους είδα, συζητήσαμε. Πρόκειται για πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το τι κάνουμε στον τομέα της γεωργικής πολιτικής, για τις εφαρμογές, για την συνέχεια που θα δώσουν αυτές οι αποφάσεις μας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα όμως να πω κάτι στον εκπρόσωπο της Επιτροπής και σε όλους όσους είναι σήμερα εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για μας για να κάνουμε αυτό που λέμε, αλλά κυρίως για τους γεωργούς, για τους αγρότες, για όλους αυτούς οι οποίοι περιμένουν αυτές τις αποφάσεις, γιατί είναι σημαντικές για την καθημερινή του ζωή. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε ακόμα κάποιες μέρες να ολοκληρωθεί το κείμενο, κατόπιν να μεταφραστεί αλλά πρέπει πριν το τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία και να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο ε, θα ήθελα να το προσέξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Το τελικό λόγο έχει ο Αλμπερντές. Ευχαριστώ για όλους όσους πήραν το λόγο, για όλα όσα είπατε. Κοιτάξτε, η κατάσταση δεν είναι απλή. Γιατί Πρέπει τώρα να ολοκληρωθεί το κείμενο. Πολλά εξαρτώνται από αυτά που θα υποβληθούν σαν προτάσεις. Ελίζαμπετ, εγώ πολύ θα ήθελα να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Ελπίζω πάντως να μπορέσουμε να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο όπως είπα αρχικά. Άκουσα πολύ προσεκτικά από αυτά που μου είπατε. Πρέπει να συνεργαστούμε διαπιστώνω από αυτά που μου είπατε ότι πρέπει να συνεργαστώ με όλους εσάς, τους κοιόδης εισηγητές, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να μπορέσουν και οι αγρότες τα επόμενα χρόνια να βρεθούν σε μια καλύτερη κατάσταση και να μπορέσουν να ε, χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια τα οποία είναι για, την, ε, είναι για δική τους χρήση. Κοιτώντας πιο προσεκτικά τα διάφορα μέτρα και τις προτάσεις για τη μεταβατική περίοδο, θα ήθελα να πω εδώ στην Επιτροπή ότι θα πρέπει εδώ να διασφαλίσουμε τις επενδύσεις, αυτές που έχουν ξεκινήσει, αυτές που είναι εν εξελίξη. Σε καμία περίπτωση το 2014 δεν μπορούμε να διακόψουμε επενδύσεις που είναι προγραμματισμένες ή που έχουν ξεκινήσει. Αυτό δεν γίνεται εν μέσω μιας ε, κρίσης σαν και αυτή που περνάει η Ευρώπη σήμερα. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις ε, θέσεις της όσον αφορά την ε, ανάγκη για έναν μεταβατικό κανονισμό. Εγώ χαίρομαι για αυτό που άκουσα από την Επιτροπή ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητο. Ελπίζω θα μπορέσουμε να βρούμε ένα συμβιβασμό. Σίγουρα το κείμενο το οποίο θα σας υποβάλω θα υποστεί τροποποιήσεις και θα συμπεριλάβω τροπολογίες. Θα εξεταστούν έτσι και αλλιώς οι τροπολογίες το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά νομίζω ότι μπορούμε να το τηρήσουμε, είναι ρεαλιστικό. Άκουσα επίσης ε, και τον γειτονά μου, ο οποίος μου είπε ότι ενδεχομένως μπορούμε να συντομεύσουμε λίγο κάποιες διαδικασίες. Κοιτάξτε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να τηρήσουμε όλες τις δυνατότητες που μέχρι τώρα υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αγρότες και αυτό μέχρι το 2016 δεν υπάρχει λόγος να δυσκολέψουμε την κατάσταση για τους γεωργούς το 2014. Όσον αφορά τουλάχιστον τις άμεσες πληρωμές, νομίζω ότι δεν πρέπει τίποτα να αλλάξει για το 2014. Δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα για το 2014. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις προτάσεις σας και φυσικά πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να συνεχιστεί. Πολύ καλά, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 8. Διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις μειονακτικές περιοχές και στις εξάχως απόκεντρες περιοχές μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος. Εισηγητής ο Χέρμπερτ Ντόρφμαν. Συνάδελφοι, αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές οι μειονεκτικές περιοχές και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές μετά το τέλος των ποσοστώσεων του γάλακτος. Είναι δύσκολες οι συνθήκες παραγωγής γάλακτος στις περιοχές αυτές, γι' αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή εμείς από πλευράς μας, ώστε το τέλος των ποσοστώσεων να μην διακυβεύσει την κτηνοτροφία και την αγροτική ανάπτυξη στις περιοχές. Να δώσω αμέσως το λόγο λοιπόν στο Χέρμπερτ για να μας κάνει την παρουσίασή του έχει ζητήσει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό και δεν θέλω να κατευθυνθούμε προς λανθασμένη κατεύθυνση. Όσον αφορά την οργάνωση της αγοράς δεν χρειάζεται κανονισμός. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν χρειαζόμαστε μεταβατική ρύθμιση για την οργάνωση της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση αυτή. Όπως είπε ο Πρόεδρος, είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό της παραγωγής γάλακτος σε μειονεκτικές περιοχές, σε απόκεντρες περιοχές, κυρίως μετά τη λήξη των ποσοστώσεων του γάλακτος. Από γνωρίζουμε υπάρχουν ε, περιοχές ορεινές, απομακρυσμένες όπου οι δυσκολίες συνεχίζουν να είναι μεγάλες, το κόστος της παραγωγής γάλατος συνεχίζει να είναι υψηλό και οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που δίνονται σε κάποιες άλλες περιοχές μέσω της απελευθέρωσης είναι κάτι που δεν ισχύει σε κάποιες απομακρυσμένες ε, και ορεινές περιοχές. Υπάρχουν περιφέρειες που δεν έχουν και άλλες εναλλακτικέ λύσεις για την παραγωγή. Παραδείγματο χάρη για παραγωγή ίνου. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν καμία δυνατότητα εναλλακτικής παραγωγής σε σχέση με την παραγωγή γάλακτος. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και θα πρέπει βεβαίως να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις. Δεν καταφέραμε βεβαίως μέχρι τώρα όσον αφορά την κοινή οργάνωση της αγοράς να συμφωνήσουμε σε ένα νέο κανονισμό. Εγώ έχω επεξεργαστεί το θέμα αυτό. Βεβαίως πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή και θα ξεκινήσω με τον πρώτο πυλώνα. Είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μέχρι τώρα υπάρχουν κράτη-μέλη που βεβαίως ε, έχουν από καιρό ε, χαρακτηρίσει κάποιες από τις περιοχές τους σε μειονακτικές, απομακρυσμένες, πολύ απομακρυσμένες, ορεινές περιοχές, περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα δεν ε, έχουν επωφεληθεί και οι οποίες έχουν δει την κατάστασή τους να επιδεινώνεται. Αυτό που σήμερα μπορούμε να πούμε είναι ότι πρέπει να τεθούν νέοι στόχοι εσωτερικής σύγκλησης. Υπάρχουν σαφώς κρατημέλη τα οποία δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες ε, επιδοτήσεων και στήριξης για αυτές τις περιοχές. Δεύτερες δεύτερη κατηγορία αν θέλετε. Υπάρχουν ε, σήμερα δυνατότητες ε, τις οποίες χρησιμοποιούν κάποια κράτη-μέλη, ειδικά προγράμματα τα οποία σε κάποιες περιφέρειες έχουν χρησιμοποιηθεί για την προστασία της παραγωγής ε, γάλακτος σε κάποιες ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Αλλά σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές ξέρετε ότι οι επενδύσεις είναι δαπανηρές, είναι πιο δαπανηρές, η πρόσβαση είναι δύσκολη, η κατασκευή είναι δαπανηρή και συγκεκριμένα εδώ θα πρέπει να στηρίξουμε τους ε, συγκεκριμένους παραγωγούς για να μπορέσουν να βρεθούν στο επίπεδο και να έχουν ίδιες δυνατότητες με άλλους. Σε πολλές ορεινές περιοχές το πρόβλημα της μεταφοράς του γάλακτος στις μονάδες επεξεργασίας είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα και οι ποσοστώσεις και η λήξη των ποσοστώσεων θα επιδεινώσουν την κατάσταση αυτών των περιοχών όσον αφορά την μεταφορά του γάλακτος στις μονάδες επεξεργασίας. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τη δυνατότητα κάποιας κρατικής επιχορήγησης έτσι ώστε να εξισορροπηθεί, να εξουδετερωθεί αυτό το επιπλέον μειονέκτημα το οποίο θα προκύψει μετά τη λήξη των ποσοστώσεων. Θεωρώ επίσης ότι σε κάποιες ε, ορεινές περιοχές ιδιαίτερα όταν ε, γίνεται επιτόπου η επεξεργασία ή όταν υπάρχει παράλληλα και τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή αυτή, να δημιουργήσουμε αγορές για τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα, τοπικές αγορές και να στηρίξουμε αυτές τις δυνατότητες ε, επεξεργασίας και διάθεσης σε αυτές τις τοπικές αγορές. Νομίζω πραγματικά όμως ότι όπως έχει σήμερα η οργάνωση των αγορών και οι προτάσεις ε, για κάποιες ε, τροποποιήσεις. Αυτό δεν φάνηκε βεβαίως ε, στον τριβερή διάλογο, αλλά νομίζω ότι εδώ στην Επιτροπή μας μπορούμε να επεξεργαστούμε τέτοιες προτάσεις μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα για τις μονάδες επεξεργασίας, μονάδες διάθεσης στην αγορά, Αναφέρομαι εδώ ιδιαίτερα σε κάποιες ε, δυνατότητες βελτίωσης ε, της επεξεργασίας τοπικών προϊόντων, διάθεσης στις τοπικές αγορές. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις δυνατότητες και να στηρίξουμε λογικές ε, προτάσεις έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις μειονεκτούσες περιοχές, τις ορεινές περιοχές. Αυτά είναι τα πρώτα σημεία τα οποία σκέφτηκα και επεξεργάστηκα. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας. Θέλω να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων. Μπορείτε να μου τις υποβάλλετε γραπτά τις επόμενες ημέρες. Χρονοδιάγραμμα όπως και ο Άλμπερντες, εγώ θα ήθελα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές να προετοιμάσω το κείμενό μου και να συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή την έκθεση. Ο Επίτροπος έχει οργανώσει μία ημερίδα με θέμα την παραγωγή γάλακτος. Θα ήταν λοιπόν λογικό νομίζω αν εμείς είχαμε ήδη τοποθετηθεί, είχαμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε μια πιο εμπεριστατωμένη πρόταση. Είμαι στη διάθεσή σας, αλλά περιμένω με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία τις προτάσεις σας. Ευχαριστώ, Χέρβερτ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έχουν ζητήσει το λόγο διάφοροι συνάδελφοι. Η Ελίζαμπεθ πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόφμαν για την πρωτοβουλία του. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον θέμα και είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν λύσεις για αυτές τις περιοχές που πραγματικά σήμερα έχουν σοβαρές ε, δυσκολίες και σε ένα τομέα όπως το γάλα που είναι εξαιρετικά ευαίσθητος. Θα πρέπει εδώ λοιπόν πραγματικά να παίξουμε το ρόλο μας και όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου και όσον αφορά αυτές τις συγκεκριμένες παραγωγές στις ορεινές περιοχές, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να προτείνουμε ειδικέ και συγκεκριμένες λύσεις Βεβαίως και οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις για τις περιοχές αυτές έχουν αντιμετωπιστεί από πλευράς της Επιτροπής με έναν τρόπο που δεν είναι ικανοποιητικός. Κάθε φορά αμφισβητείται αυτός ο τομέας. Για μας είναι πραγματικά παράλογο να μην μπορούμε να βρούμε έναν ε, αποτελεσματικό τρόπο στήριξη με άσεμε πληρωμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτές τις περιοχές, τις συγκεκριμένες ορεινέ περιοχές, να βρεθούν συγκεκριμένες λύσεις. Υπάρχει υψηλό κόστος παραγωγής, η πρόσβαση είναι δύσκολη, η μεταφορά είναι δύσκολη. Γι' αυτό ακριβώς και θα πρέπει να στηρίξουμε με ειδικά μέτρα τις ε, περιοχές αυτές και πραγματικά στηρίζω τις προτάσεις του εισηγητή ιδιαίτερα όταν λέει ότι πρέπει να βελτιώσουμε την πρόσβαση και ότι κάποια ειδικά προϊόντα με προστιθέμενη αξία θα πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα. Ο καταναλωτής βεβαίως σήμερα γνωρίζει και ζητάει αυτήν την ε, ειδική ποιότητα αυτών των προϊόντων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι σε αυτές τις περιοχές η γεωργική παραγωγή είναι μια παραγωγή η οποία στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης σε αυτές τις ε, περιοχές εξαρτώνται από πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και εδώ πρέπει πραγματικά να συνειδητοποιήσουμε τη στρατηγική σημασία των μέτρων που πρέπει να πάρουμε για την στήριξη αυτών των παραγωγών. Συμφωνώ και εγώ ότι η διάθεση στην αγορά, η διανομή, η στήριξη των τοπικών αγορών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσω των συνεταιρισμών, μέσω κοινών πρωτοβουλειών, παραγωγών και γεωργών και όλα αυτά θα πρέπει να συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα παραμείνουν ζωντανές αυτές οι περιοχές και στο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να δραστηριοποιηθούμε και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Ντόρφμαν για την πρωτοβουλία του. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντόρφμα μας έδωσε πολύ καλές ιδέες. Μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά νομίζω κάτι ξέχασε. Το ότι στις διαπραγματεύσεις για το πακέτο του γάλακτος ήταν σαφές στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής ότι το Συμβούλιο, μάλλον η Επιτροπή, δεν έχει αντιμετωπίσει το θέμα της, του προσανατολισμού αυτής της αγοράς, όπως ακριβώς έκαναν και με τον Ίνο. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι πώς θα μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με τα κονδύλια που διαθέτουμε. Κάθε φορά βλέπουμε, παραδείγματο χάρη στη Γερμανία, όταν μιλάμε για τις ορεινές περιοχές, αλλά όχι μόνο τις ορεινές περιοχές, κίνηση, η κατεύθυνση αν θέλετε να είναι από τον νότο προς το βορρά να μεταφέρονται τα προϊόντα και να στηρίζουμε περιοχές μειονεκτικές άσχετα με το που παράγεται με τον καλύτερο και το πιο οικονομικό τρόπο ένα προϊόν. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τις ε, ορεινές περιοχές της Άλπης παραδείγματο χάρη, στη Γερμανία έχουμε πολλές άλλες περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις παραγωγής. Πρόκειται λοιπόν εδώ για ένα πάρα πολύ ακριβό δαπανηρό πρόγραμμα και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Στις συζητήσεις που έχουμε με την Επιτροπή που θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο και την ημερίδα που θα οργανωθεί για το θέμα αυτό, Όπως είπατε κύριε Ντόρφμαν, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους και να πούμε ότι εδώ πρέπει να κατανείμουμε αυτά τα συγκεκριμένα κονδύλια στους παραγωγούς και στους γεωργούς που βρίσκονται σε αυτές τις ορεινές περιοχές. Υπάρχει και άλλη δυνατότητα, μπορεί να δοθεί μια άλλη κατεύθυνση στην αγορά του γάλατος και ενδεχομένως αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε Πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει και αυτό να μπει στη συζήτηση. Πώς κατανέμονται αυτά τα κονδύλια. Και αυτό αποκοινούμε τις δικές σας προτάσεις. Ευχαριστώ Μάρτιν, ο κύριος Άγνιο και μετά η Μπρίτα Ρέμερς. Σε όλη την Ευρώπη και στις Βρετανικές νήσους έχουμε πάντοτε αυτό το πρόβλημα, το δίλημα, όπου άτομα προσπαθούν να έχουν γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις με πάρα πολύ δυσμενείς περιπτώσεις, διότι η αγορά έχει απομακρυνθεί από αυτούς δεν μπορούν να αναπτυχθούν, ίσως ε, γιατί ίσως το έδαφος δεν είναι αρκετά καλό, δεν μπορούν να έχουν δασοκομεία, ε, χρειάζεται να παίρνουν τρόφιμα συμπυκνωμένα, σημαίνει ότι ε, φορτηγά, μεγάλα φορτηγά περνάνε από κακούς δρόμους και πρέπει το γάλα να συλλέγεται τρεις ή τέσσερις φορές τη βδομάδα. Αν πείτε, ας ξοδέψουμε περισσότερα χρήματα στον τομέα αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ναι, ας έχουμε ένα ταμείο να επιτρέψουμε σε αυτούς τους τα άτομα να συνταξιδοτηθούν με αξιοπρέπεια ή να περάσουν ίσως σε άλλους τομείς, να περάσουν σε βοηδή, σε πρόβατα ε, και υπάρχει και επίσης αυτή η να περασουν ισως σε αλλους τομεις να περασουν σε βοηθη σε προβατα και υπαρχει και επισης αυτη η κτηνοτροφια είναι καλή για αυτές τις περιοχές να μπορέσουν, ε, βλέπει κανείς, να πουλήσει, να, να αποθηκεύσει στο τέλος του Αυγούστου, ενώ υπάρχει ακόμα χορτάρι. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τα πράγματα από διαφορετική ε, μορφή και πλευρά. Η γαλακτοκομική εκμετάλλευση δεν είναι αυτό που ήταν πριν από 60 χρόνια, τα βοσκοτόπια και αυτά. Δεν μπορούμε να ζούμε στο παρελθόν. Ευχαριστώ Άγνιο, Μπρίτα και μετά Σεκεριέσκη. Yeah, Ευχαριστώ οι ορεινές περιοχές που έχουν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κτηνοτροφία, παραγωγή γάλατος, σίγουρα στοιχίζουν πολύ περισσότερο. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την παραγωγή, όχι μόνο σαν ε, μια παραγωγή που κοστίζει παραπάνω, αλλά σε σχέση με την ανάπτυξη τη γενικότερη της ε, περιοχής αυτής, της υπαίθρου, της περιφέρειας, αν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις και αν υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρξει ανάπτυξη της ε, εργασίας, της απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα προγράμματα αυτά με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως ε, τα... η παραγωγή αυτή δεν είναι μια παραγωγή οικονομική. Το θέμα είναι τι εναλλακτικέ λύσεις έχουν αυτές οι περιοχές, τι μοντέλο διαφορετικό μπορούμε να προτείνουμε και αν δούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο θα πρέπει πραγματικά να στηρίξουμε με προγράμματα και θα ήθελα αυτές οι προτάσεις να στηρίζονται και στους τρεις πυλώνες και στην ανάπτυξη της πέτρου και στην ε, γεωργική παραγωγή και βεβαίως στον κοινωνικό παράγοντα. Και να κοιτάξουμε βεβαίως και τις ε, αρνητικές ε, επιπτώσεις. Να μην υπάρξει παραδείγματος χάρη διακριτική προτιμησιακή χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων. Υπάρχουν περιοχές που ναι μεν δεν καλύπτονται από αυτά τα κριτήρια, δεν μπορούν δηλαδή να υποφεληθούν από αυτή τη χρηματοδότηση, από αυτά τα προγράμματα. Είναι όμως εξαιρετικά μειονεκτικές περιοχές. Ας κοιτάξουμε λοιπόν αυτή η επιλογή να μην έχει αρνητικέ συνέπειες σε άλλες περιοχές που δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτά τα προγράμματα. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε τα διαρθρωτικά προβλήματα αυτών των περιοχών, των ορεινών, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου η γεωργική παραγωγή, η αγροτική ανάπτυξη έχει άμεση σχέση με τον τουρισμό. Είναι πολλές φορές ε, πάρα πολύ μεγάλη η σχέση που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές μεταξύ του τουρισμού, της παραγωγής και της ανάπτυξης του υπέρχου. Ευχαριστώ Μπρίτα. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να βρούμε και κάποια οικονομικά ωφέλη. Συνεχίζω από αυτά που είπε ο κύριος Άγνιου. Ακόμα και αν ισχύουν αυτά τα οποία είπατε, θα πρέπει να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στους ανθρώπους στις ορεινές ε, περιοχές εκ των προτέρων. Συμφωνώ όμως με τους περισσότερους από τους ε, και θεωρώ ότι το θέμα αυτό, η γαλακτοπαραγωγή εν γέννη και ε, το τι θα γίνει όταν θα εκπνεύσουν οι ποσοστώσεις ε, είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει στην νομοθεσία για το γάλα και πρέπει απλώς να διευκρινίσουμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ καλό ότι υπάρχει η έκθεση αυτή αυτή τη στιγμή και το γεγονός ότι το θέμα αυτό επισημαίνεται καταλήλως. Η γαλακτοπαραγωγή στις ορεινές περιοχές, διότι ε, σε αυτή την περίπτωση αναφερόμαστε κυρίως ε, σε μικρές εκμεταλλεύσεις οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν έναν τρόπο ζωής συγκεκριμένο και να μπορούν να επιβιώσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε αυτό στην έκθεση, να έχουμε τη σαφή σχέση ε, με την νομοθεσία για το γάλα, διότι πρέπει να αποφύγουμε και κάποιες συγχύσεις. Ε, όλοι λένε ότι η απόφαση είναι πλέον ηλυμένη και απομένει να εφαρμοστεί. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε εδώ και θα πρέπει να το αποδείξουμε. Το συζητάμε αυτό τώρα που ολοκληρώνουμε και τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση. Θα μπορούσαμε κάποιος να πει λοιπόν ότι έχουμε καθυστερήσει, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Διότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, υπάρχει δυνατότητα να βρούμε κάτι στο δεύτερο πυλώνα για να στηρίξουμε το συγκεκριμένο τομέα. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να αλλάξουμε και λίγο νοοτροπία όσον αφορά τη στήριξη ε, αυτών των ανθρώπων από εθνικές πηγές. Η παραγωγή γάλακτος σε αυτές τις τόσο μικρές εκμεταλλεύσεις ελάχιστα επηρεάζει την κατάσταση της αγοράς, διότι τις περισσότερες φορές πρόκειται απλώς ε, για τοπική παραγωγή που καλύπτει την ανάγκη του τοπικού πληθυσμού και ίσως και κάποιους τουρίστες. Η ε, επιρροή λοιπόν που έχει στην αγορά του γάλακτος είναι ελάχιστη και θα μπορούσαμε ίσως να προβλέψουμε και κάποια στήριξη από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Ε, πάντα βέβαια με τη δέουσα εποπτεία, διότι θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εποπτεύει τα πάντα και δεν θα πρέπει φυσικά να ανοίξουμε και την ε, ε, δυνατότητα να ε, υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να δοθεί μια κάποια μορφή στήριξη είτε για τη μεταφορά είτε για την επεξεργασία στη συνέχεια και τη μεταποίηση του γάλακτος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να επιβιώσει και αυτή η τόσο μικρή κλίμακα παραγωγή. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι αυτές οι ορεινές περιοχές ε, είναι πάρα πολύ ευέλικτες, υπάρχει τουρισμός, ε, τοπικά προϊόντα και είναι διαφορετική η προσέγγιση προς την παραγωγή και προς τη ζωή, διότι η παραγωγή στις ορεινές περιοχές είναι μια έκφραση ζωής, πολιτισμού αν θέλετε και θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και χαίρομαι ιδιαίτερα που συζητάμε τα συγκεκριμένα θέματα σήμερα και θα τα συζητήσουμε και στο μέλλον. Ιδίω και το θέμα της οικονομική παραγωγής διότι εκεί θα πρέπει να καλύψουμε και τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ε, και αυτές τις εκμεταλλεύσεις σήμερα. Πριν ολοκληρώσουμε φυσικά και τη συζήτηση για τον ε, προϋπολογισμό της ΚΑΠ και τη μεταρρύθμιση, ο Λουίς Καπουλασάντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια μικρή παρέμβαση και για, ε, προσωπικά και για τον Λούις Παλουράσιος που είναι ο σκιώδης εισηγητής αλλά λόγω πολιτικών υποχρεώσεων εθνικών δεν μπορεί να βρεθεί εδώ σήμερα. Μιλάω λοιπόν προσωπικά και για αυτόν. Εγώ προσωπικά Πάντοτε ανέφερα τη μεγάλη μου ανησυχία σχετικά με τις λύσεις που προτείνονται για τον γαλακτοκομικό τομέα, ακόμα και αυτό που αποφασίστηκε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ΚΑΠΑ για τις, ε, για τις ορεινές περιοχές, για τις μειονεκτικές περιοχές και τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Έχω πάει στην ε, περιφέρεια του Herbert Dorfman ε, και με καθησυχάζει το ότι αυτός είναι ο εισηγητής του φακέλου αυτού, διότι κατανοεί πολύ καλά τα προβλήματα ε, που θέτει ο τομέας. Οι Ασόρες, τα νησιά που βρίσκονται στα μέσα του Ατλαντικού, τα νησιά παράγουν εν τρίτον του γάλακτος της χώρας μου και αυτά τα νησιά δεν έχουν άλλη οικονομική και κοινωνική εναλλακτική λύση. Το μόνο που μπορούν είναι να εκμεταλλεύονται το έδαφος που έχουν. Όταν λοιπόν διαπιστώνουμε ότι τα εναλλακτικά, τα μέτρα ε, τείνουν ε, να ε, μειώσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις των, των ποσοστώσεων γάλακτος, όλα αυτά είναι ανησυχητικά ότι θα τελειώσουν. Περιμένω την μελέτη που θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο που παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέτρα που θα μπορέσουν να μετριάσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στις περιοχές οι οποίες είναι οι πιο πτωχές, οι πιο μειονεκτικές, οι οποίες ε, καλύπτονται λιγότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πώς αυτές τις επιπτώσεις ε, θα, θα μειωθούν αυτές οι επιπτώσεις, πώς θα περιοριστούν και θα περιοριστεί επίσης ε, και η μετανάστευση από αυτές τις περιοχές και η έξοδος από τις αγροτικές περιοχές. Ελπίζω να μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Jim και μετά ο George Lyon. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο γαλακτοκομικός κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας ενώ προχωρούμε ε, και ενώ και όταν ε, οι ποσοστώσεις θα εξαλειφθούν και όταν θα υπάρξει ένα νέο σύστημα που θα ισχύσει. Εγώ θυμάμαι πώς ήταν ε, η ζωή πριν από τις ποσοστώσεις και μπορώ να θυμηθώ ότι τότε εισχολούμουν με την πολιτική και ήμουν μέλος ε, ενώσεων και ερχόντουσαν διάφοροι αγρότες και μου λέγανε πώς οι θα επηρεάσουν την ε, γαλακτοκομική παραγωγή. Ε, επειδή κάτι όμως τώρα υπάρχει τόσο πολύ καιρό και θα αλλάξει, δεν σημαίνει απαρατήτως ότι, ότι αυτό θα είναι κακό μακροπρόθεσμα για τον κλάδο. Πέρσι αυτήν την εποχή πήγαμε ε, στην περιφέρεια του κυρίου Ντόρφαν και η, Ελίζα, Ελίζαμπεθ ε, οργάνωσε πάρα πολύ καλό, καλή επίσκεψη και είδαμε τα προβλήματα της περιοχής αυτής και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν άλλες περιφέρειες στην Ευρώπη και στην δική μου περιοχή και ο κύριος Άγνιο έχει δίκιο, υπάρχουν μερικά ε, μέρη, μερικές περιοχές που είναι καλύτερες για πρόβατα, για, για κτηνοτροφία κλπ. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε ε, σε σχέση με την κατάσταση, ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι αγροτικό πρόβλημα ή οικοκοινωνικό πρόβλημα. Πώς το αντιμετωπίζουμε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις ε, ε, μπορώ να καταλάβω ε, ακόμα και τον κύριο Ντόρτμαν που μίλησε γερμανικά που έχουμε τα όσα λέει η Μαριαν Φίσερ Μπόουλ αλλά όταν το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε να εξαλείψει τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις είχα την ευθύνη ε, να είμαι εισηγητής για το γαλακτοκομικό πακέτο. Και είχαμε ένα πακέτο αρκετά προσεκτικό, εξισορροπημένο, ελπίζοντας ότι το γαλακτοκομικό πακέτο ε, θα είναι ικανοποιητικό, αλλά υπάρχει αρκετή προστασία για το μέλλον το Σεπτέμβριο η συζήτηση υψηλού επίπεδου, παρόλο που δεν ξέρουμε τι θα συζητήσουμε, θα είναι όμως πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και αυτό ε, που θα πρέπει να γίνει στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι ότι ποτέ, ποτέ η Κομισιόν δεν θα πρέπει να μπορεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να μας λέει ότι τίποτα δεν ε, πάει άσχημα στον γαλακτικό κομικό τομέα όταν Ξέρουμε ότι για δύο χρόνια προτού δράσει η Κομισιόν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Πώς θα γίνει αυτή η ομαλή προσγείωση. Βλέπουμε πώς έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και πώς οι γαλακτοκόμοι περιμένουν κάτι καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι με το πακέτο το γαλακτοκομικό, με τη μεταρρύθμιση της Ούτε το Συμβούλιο ούτε η Κομισιό έχουν την πρόθεση νομίζω να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν ε, τους ανθρώπους σε αυτές τις τόσο ευάλωτες ε, περιοχές. Ε, βεβαίως αυτό που δεν θέλω, δεν θέλω κανείς, κανείς από εμά δεν θέλει να δει το τίμημα που θα πρέπει να πληρωθεί για να παραμείνουν οι περιοχές ως έχουν. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε όμως μια ευθύνη απέναντι τους. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω ε, τι θα πρέπει να γίνει, πώς θα μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα, αλλά θα υπάρξει ένα μαζικό πρόβλημα αν ε, συνεχίσουμε να έχουμε την ερημοποίηση αυτών των περιοχών. Αυτό θα είναι μεγάλη δυστυχία μακροπρόθεσμα, μεγάλη κακοτυχία. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε εδώ και ήρθε η ώρα να κάνει ο κύριος Ντόρφμαν αυτήν την εισήγηση. Δεν ξέρω αν θα δημιουργηθούν μεγαλύτερες δυσκολίες για το γαλακτοκομικό τομέα σε αυτές τις ορεινές περιοχές, τις μειονεκτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Αλλά δεν ξέρω ποια λύση θα μπορούμε να βρούμε. Ευχαριστώ, Τζιμ. Ο Τζορτ Λάιον και μετά η κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εκ μέρου ε, του συναδέλφου Ρίκα Μπάκεν, είναι ο σκιώδη ηγητή των Φιλελευθέρων ε, για το θέμα αυτό και ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα. Είχε κάποια άλλη πολιτική δέσμευση και δεν μπορούσε να είναι παρούσα εδώ σήμερα από την ε, Φιλανδία και να είναι γέρο στη συνεδρίαση. Εγώ όταν ε, τελείωσα το σχολείο για 15-16 χρόνια άρμεγα γελάδες και γνωρίζω λίγο κάποιες από τις προκλήσεις του να προσπαθεί να κερδίσει κάποιος χρήματα από την ε, παραγωγή γάλακτος. Ε, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στη Φιλανδία με μια πολύ μικρότερη ε, περίοδο ανάπτυξης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στη Σκωτία φαίνονται ασήμαντες. Και αυτά τα θέματα ήθελε να τα θίξει η συνάδελφος η Ρίκα, ε, γιατί υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες για την παραγωγή γάλακτος σε κάποιες από αυτές τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στον αρκτικό κύκλο. Καλωσορίζει ε, το γεγονός ότι επικεντρώθηκε η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, στην δυνατότητα να υπάρχουν κάποια εργαλεία που θα μπορέσουν να διασφαλίσουν ότι θα λαμβάνουν τη στήριξη που χρειάζονται αυτές οι περιοχές και θα διατίθεται στήριξη, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό που είπε ο συνάδελφο από το UKIP, να του δώσουμε δύο δεκάρε και να του πούμε να εξαφανιστούν στα εξών συνετέθησαν. Αυτό είναι παράλογο από πολιτική σκοπιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει παραγωγή γάλακτο στη Φιλανδία καθόλου. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες ώστε να υπάρχει συνεχή στήριξη και για το μέλλον, διότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει η παραγωγή σε ε, αυτές τις περιοχές που είναι τόσο σημαντικό όχι μόνο από πλευράς παραγωγής αλλά κυρίως από κοινωνική σκοπιά ώστε να διασφαλίσουμε και την ε, επιβίωσή τους και την παραμονή τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το να παραμείνει η παραγωγή γάλακτος διότι είναι πολύ ε, ευμετάβλητες οι τιμές ε, και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να βγάζουν τα προστοζήν θα μεταφέρονται σε άλλες περιοχές ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδείξουμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η παραγωγή γάλακτος σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στις περιοχές που μπορούν να είναι πραγματικά ανταγωνιστικές και μπορούν να παράγουν γάλα χωρίς στήριξη στο μέλλον. Ευχαριστώ η Μάριαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εν είδη εισαγωγή να σας πω ότι νιώθω λίγο κτηνοτρόφο αυτή την ε, επιτροπή, διότι νόμιζα ότι ε, είχαμε τελειώσει την περασμένη εβδομάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται μόλις αρχίζουμε. Μέτρα για το πολιτευστημο δημοσιονομικό πλαίσιο, διάμεσα μέτρα, μεταβατικά μέτρα και η έκθεση αυτή. Ζήτησα το λόγο γιατί πήγα επιτόπου ε, στην αποστολή που μας κάλεσαν η Ελίζαμπεθ και ο Χέρμπερτ και πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε και να φροντίσουμε επενδύσουμε σε αυτές τις περιοχές. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να βοηθήσουμε το Χέρμπερτ με την έκθεση το υποστηρίζω. Οπότε ξέρετε εγώ κατάγομαι από την Ιρλανδία που είναι ανταγωνιστική στον τομέα αυτό και δεν νομίζω ότι ο Άγνιου το είπε ε, αρνητικά, το είπε από σεβασμό ότι θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν αυτοί οι κτηνοτρόφοι. Εάν το κάνουμε αυτό, ε, θα πρέπει σε τρία με πέντε χρόνια να αρχίσουμε να πληρώνουμε κτηνοτρόφους, να αρχίσουν και πάλι να παράγουν γάλα. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν και ίσως εάν συζητήσουμε το θέμα αυτό στην κοινή αγροτική πολιτική θα ε, μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα στοιχεία. Ε, πρέπει να στηρίξουμε το Χέρμπερτ για την πρωτοβουλία αυτή, είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να ακούσουμε και την άποψη των κτηνοτρόφων. Τι άποψη έχουν αυτοί χρειάζεται να παραμείνει ζωντανή ε, η παραγωγή σε αυτές τις περιοχές και οτιδήποτε διατηρήσει ζωντανές αυτές τις περιοχές ε, και την παραγωγή γάλακτος θα βοηθήσει. Θέλω λοιπόν να ε, προωθήσουμε την έκθεση αυτή και θα την υποστηρίξω φυσικά εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Άγνιου θέλει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επανέλθω, γιατί νομίζω ότι ο κύριο Λάιον ήταν άδικο. Είπα απλώ να συνταξιοθετηθούν με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα του δώσουμε δύο δεκάρε σε καμία περίπτωση. Και είπα ότι κάποιοι από αυτού του ανθρώπου θα μπορούσαν να παραμείνουν στις παραγωγέ του, στι εκμεταλλεύσει του και να ε, χρησιμοποιήσουν την εκμετάλλευση για πολύ πολύ καλύτερη παραγωγή. Πολύ καλά, τα διευκρινίσαμε και αυτά. Ευχαριστώ, Άλμπερτ Τέστορα. Εγώ ήθελα να πω στον ε, συνάδελφο τον κύριο Άγνιο ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να εγκατασταθεί και να διαρκέσει σε αυτές τις περιοχές αν παράγει γάλα. Αν γνωρίζει κανείς ε, το τι κάνουν η Ελίζαμπετ, παραδείγματος χάρη, σε κάποιες περιοχές, το τι ρόλο και άλλοι, ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο στο νότιο Τυρόλο παραδείγματος χάρη Ελάτε να δείτε πώς ε, παράγονται διάφορα προϊόντα. Οι δυσκολίες είναι πολλές, οι εποχές ε, δύσκολες και καλό θα ήταν κάποιοι από εμά να πάνε να κάνουν ε, μια μικρή άσκηση, μια μικρή μαθητεία σε κάποιες από αυτές τις ε, συγκεκριμένες περιοχές θα δείτε πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση από αυτή που επικρατεί σε μία παιδιάδα, σε μία άλλη έφορη περιοχή. Πώς εργάζονται αυτοί οι γεωργοί πολλές φορές με όλη τους την οικογένεια και πόσο διαφορετική είναι η παραγωγή και ο τρόπος παραγωγής. Ευχαριστώ πολύ γιατί ξέρω ότι πολλοί συμφωνούν και γνωρίζουν αυτή την κατάσταση. Τώρα, στη Φιλανδία που υπάρχουν ορεινές περιοχές. Ε, αν αρχίσουμε τώρα βέβαια μια συζήτηση για το πού είναι πιο δύσκολη η παραγωγή σε νησιά, σε ορεινά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συμπεριλάβουμε πραγματικά σε αυτή την κατηγορία όλες αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, περιοχές μειονεκτικές, απόμακρες, ορεινές, που συνεχίζουν όμως να παράγουν ε, γάλα. Και όταν βλέπω ότι σε αυτές τις επειδή υπάρχει παράδοση, ιστορική παράδοση για την παραγωγή αυτή, συνεχίζουν κάποιοι να παράγουν με μια στήριξη 16 ευρώ, ενώ στην Λομβαρδία παραδείγματο χάρη το αντίστοιχο ποσό είναι 60, καταλαβαίνετε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε αυτή η παραδοσιακή παραγωγή, αυτή η παραδοσιακή ζωή και ανάπτυξη αυτών των περιοχών να την στηρίξουμε. Ξέρω πολύ καλά την περιοχή του Νότιου Τυρόλου και στην δική μας ομάδα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε η λύση που θα υιοθετηθεί να είναι λογική. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν Όσλιν και μετά θα δώσουμε το λόγο στο Χέρμπερτ. Μάρτιν. Θα ήθελα να πω ότι το θέμα δεν είναι τι θα κατανείμουμε σε αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για ένα μικρό ποσό που θα πάει από το δεύτερο πυλώνα. Και έτσι κι αλλιώς έχει μειωθεί το ποσό αυτό που συνολικά ε, θα στηρίξει την παραγωγή γάλατος. Από πού λοιπόν θα προέρχεται αυτό το επιπλέον περιεχόν, από κάπου αλλού θα βγει. Θέλω να σας πω και ελπίζω, Χέρμπερτ, να πετύχεις αυτό που θέλεις, αλλά το θέμα είναι να ληφθούν και μέτρα της αγοράς, έτσι ώστε η κατεύθυνση που θα δοθεί σε αυτή την παραγωγή να είναι με προοπτικές. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το πόσα ευρώ παραπάνω θα δοθούν, θα κατανεμηθούν και αν θα φύγουν από το δεύτερο πυλώνα ή αν θα είναι... Ε, αν θα πρόκειται για συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, συγητής. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις ακούστηκαν και ευχαριστώ όλους. Εγώ τα έχω σημειώσει όλα όσα είπατε. Να πω στον κύριο Όσλινγκ. Στις ορεινές περιοχές υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες και προβλήματα. Εάν θέλει κάποιος να πάρει μέτρα για την οργάνωση της αγοράς, όπως είπες, σε αυτή την περίπτωση αυτό ισχύει για όλη την παραγωγή, για όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε την παραγωγή γάλακτος στην Ευρώπη και να την κάνουμε λίγο πιο ελκυστική, σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε δυνατότητες και θα τις κατευθύνουμε στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και όχι σε αυτούς που έχουν μικρή επιφάνεια, άρα μικρή παραγωγή και συγκεκριμένες δυσκολίες. Αυτό είναι το δίλημα εδώ που έχουμε. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους για τις συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στα συγκεκριμένα μέτρα, στη συγκεκριμένη στήριξη που χρειάζονται αυτές οι περιοχές και θα πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε αυτές οι περιοχές να μπορέσουν να αποκτήσουν κάποια πλεονεκτήματα που να εξισορροπήσουν τα μειονεκτήματα που έχουν έναντι άλλων περιοχών. Δεν σας αρέσει αυτή η διατύπωση, το κάνω όμως λίγο επίτηδες. Η συνάδελφος Κέρστινγκ ε, έρχεται από μια πολύ όμορφη περιοχή. Μπορούμε όντως να πάμε να την επισκεφτούμε και στη δική μου περιοχή μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι γιατί νομίζω ότι εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν νέοι, νέα παιδιά που εργάζονται, που παράγουν και εγώ προσωπικά σας καλώ να έρθετε στην περιοχή μου για να καταλάβετε γιατί ακριβώς φαινόμενο ε, συζητάμε εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ όλους και νομίζω ότι πρέπει πολύ γρήγορα να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της μερίσιας διάταξης, διότι έχουμε ελάχιστα λεπτά και θα πρέπει στη συνέχεια να φύγουμε από την αίθουσα. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε όλοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το προσχέδιο προπολογισμού για το 2014, το οποίο αποτελεί την πραγματική έναρξη της διαδικασίας του ετήσιου προπολογισμού. Στα τέλη Ιουνίου, οι πρόεδροι των τριών ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων κατέληξαν σε συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, το οποίο επιβεβαιώνει τους περιορισμούς στον προπολογισμό που επέβαλε το Συμβούλιο το Φεβρουάριο και ε, τους οποίους υπερψηφίσαμε και εμεί την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, αγαπητοί συνάδελφοι. Στον τίτλο 2 του πολετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου που περιλαμβάνει και ε, την γεωργική πολιτική θα υπάρξουν σημαντικές περικοπές για τα επόμενα χρόνια, όπως μας εξήγησε και το Τμήμα Πολιτικής σε μια παρουσίαση που μας έκανε πριν από κάποιους μήνες. Επομένως, ο προπολογισμό για το 2014, το πρώτο έτος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα έχει περικοπές της τάξης του 5% λόγω της εφαρμογής του μηχανισμού της δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο. Το προσχέδιο προπολογισμού προβλέπει και άλλες περικοπές για τα μέτρα της αγοράς και για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ωστόσο, όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, όπως εξήγησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εδώ έχουμε και τον ε, διευθυντή, τον οποίο καλωσορίζω, τον κύριο Λόμπο, στην αρχή της προγραμματικής περίοδου χρειαζόμαστε ένα χαμηλό επίπεδο πληρωμών. Όπως λοιπόν και για τις προηγούμενες χρονιές θα πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίες πριν από την ε, ε σκαλοκαιρινές διακοπές και υπάρχει προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 22 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Να δώσω τώρα το λόγο στη συντάκτρια της ε, γνωμοδότησης, την κυρία Ντάνσιλα. Ναι, έχουμε μια καθυστέρηση ενός μηνός που μας εμπόδισε να έχουμε ένα σχέδιο. Στις 27 Ιουνίου τα τρία βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήγγυλαν ότι συμφώνησαν για ένα σχέδιο πρότασης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και εκπώνησαν για το 2014 το σχέδιο προϋπολογισμού. Όπως είπανε στον τίτλο 2 που περιλαμβάνει την κοινή αγροτική πολιτική. Αν πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συμφωνία του, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουμε μια συνολική μείωση 3,4% από 346 373,2 ευρώ. Αν πρέπει να συγκρίνουμε ε, ε, το πολιετές πλαίσιο 2007-2013 με το 2014-2020, η μείωση θα είναι μείον 11,3%. Όπως είπατε, είναι σημαντική περικοπή. Όσον αφορά ε, τον προϋπολογισμό του 2014, ε, οι πιστώσεις ε, πληρωμών ε, του τίτλου 2 μειώνονται για όλες τις κατηγορίες κατά 2,3% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013. Όπως αναφέρεται δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, γι' αυτό δεν θα μπω σε λεπτομερή ανάλυση, αλλά θα ήθελα ωστόσο να αναφέρω ότι όλοι οι αγρότες στρέφονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ε, Γεωργίας και νομίζω ότι φέτος που είναι μια, ένα μεταβατικό έτος που είναι σημαντικό για όλους τους ευρωπαϊκούς αγρότες θα είναι έτος αποφασιστικό. Νομίζω ότι αυτή η περικοπή πρέπει να συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή και πρέπει να βρούμε λύσεις μαζί βεβαίως, λύσεις μαζί ούτως ώστε να δώσουμε μια κατάλληλη απάντηση στους ανθρώπους που στρέφονται σε μας για βοήθεια, όχι για περικοπές δημοσιονομικές. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω το γεγονός ότι θα έχουμε αύριο μια συνάντηση ε, με τον εισηγητή του προϋπολογισμού και θα σας αναφέρω τις λεπτομέρειες σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020. Όπως ήδη αναφέρατε, η προθεσμία είναι 22 Ιουλίου στο μεσημέρι για τις τροπολογίες και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι στο σχέδιο αυτό έχουμε 16 σχέδια πιλωτικά 11 ε, και 6 9. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ την κυρία Ντάντσιλα. Εάν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, θα ήθελα να δώσω το λόγο. Ε, η κυρία Λούλινγκ, παρακαλώ. Μια μικρή ερώτηση μόνο. Ε, η κυρία εισηγήτρια είπε ότι θα υπάρξουν περικοπές και θα πρέπει να βρούμε λύσεις σε αυτές τις περικοπές της δημοσιονομικές. Τι μπορεί να είναι αυτές οι λύσεις όταν δεν υπάρχουν τα κονδύλια. George, εσύ να προτείνεις. Αν δεν έχουμε κρίση θα πάρουμε τα χρήματα ε, του χρόνου και θα απορροφηθούν οι περικοπές. Θα μπορούσε να είναι μια λύση και αυτή. Όχι, δεν το λέω σοβαρά, διότι πρέπει να βρούμε λύσεις. Αλλά ποια είναι η λύση. Εγώ δεν βλέπω λύση. Να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα. Ούτε και αυτό γίνεται. Είναι ότι υπάρχουν συμφωνίες. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για λύσεις και να θεωρούμε ότι ε, θα ε, δώσουμε λύσεις στους γεωργούς όταν δεν υπάρχουν. Να δώσουμε το λόγο στον Άλτο Λόγκο, μήπως μας δώσει λύσεις αυτός. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύσκολη λύση. Δεν υπάρχει και το μαγικό ελιξίριο, αλλά φυσικά θα μπορούσα να σας ε, δώσω κάποιες διευκρινήσεις για τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να περιοριστώ σε δύο ουσιαστικά σημεία σε αυτή την υπόθεση, διότι ξέρω ότι μας πιέζει και ο χρόνος. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε τη νέα κατάσταση ε, εντός της οποίας βρισκόμαστε για πρώτη φορά για το 2014 και θα ξαναβρεθούμε και ενώπιον της ίδιας κατάστασης για τα επόμενα χρόνια κυρίως για τον πρώτο πυλώνα. Η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι η πλήρης απουσία ε, περιθωρίου ευελιξίας στα επιμέρους ανώτατα όρια. Για τις γραμμές λοιπόν του Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης υπάρχει ε, μία ελάχιστη αύξηση, θα είναι μείωση, δεν μπορούμε να έχουμε μείωση, διότι η μείωση σημαίνει ότι θα μειωθεί περισσότερο η δημοσιονομική πειθαρχία. Οι δύο παράμετροι αυτές λοιπόν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία του προπολογισμού που ξεκινά σήμερα. Δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω και κάτι, κύριε Πρόεδρε, που αφορά το δεύτερο πυλώνα, την ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι πιστώσεις που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, βάση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Όσον αφορά όμως τις πιστώσεις πληρωμών, και με βάση τη συνολική συμφωνία ε, στην οποία είχαμε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κάνει μια πολύ περιορισμένη πρόταση, η οποία θα βασίζεται, και προσέξτε με εδώ, στην ε, υπόθεση ότι ο διορθωτικός προπολογισμό του 2013 θα εγκριθεί στο σύνολό του. Ξέρουμε ότι οι απαιτήσει όσον αφορά τις πληρωμές θα είναι πολύ αυξημένε διότι είναι προχωρημένα τα, παρούσα, τα παρόντα προγράμματα και φυσικά υπάρχουν και οι πρώτες πληρωμές για τα προγράμματα του 2014-2020. Οι πιστώσεις που ζητώνται για τον προπολογισμό του 2014 στο πλειονότητά τους είναι για να καλύψουμε τα προγράμματα του 2012-2013. Ε, για το 2014-2020 έχουμε προβλέψει ότι περίπου το 50% των προγραμμάτων θα εγκριθεί το 2014 και θα πρέπει να δοθούν προκαταβολές το 2014 για αυτά τα προγράμματα. Για τις πιστώσεις πληρωμών λοιπόν για την ανάπτυξη του υπαίθρου πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Λόγκο, αν και δεν μας έδωσε και αυτός καμιά λύση ή και καλά νέα, αλλά λόγω του εγωισμού των κρατών μελών δεν έχουμε και πολλές αναλλακτικές λύσεις, όπως θα θυμόμαστε όλοι. Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε και με μεγάλη σχετικά πλειοψηφία την συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεπώς έτσι έχει το πράγμα και με αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε. Δεν ξέρω αν η συνάδελφος ε, Ντάντσιλα θέλει το λόγο, αλλιώς νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε εδώ τη συζήτηση. Δεν θέλετε το λίγο, ωραία. Πέρασε συνεδρίαση. Υπενθυμίζω ότι αύριο το πρωί στις 9 θα είναι εδώ ο Λιθουανός υπουργό, γι' αυτό καλό θα ήταν να είστε όλοι παρόντες. Ευχαριστώ, καλό βράδυ.